Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να υποδεχόμαστε τον πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς και να τον καλωσορίζουμε. Αξιότιμη κυρία Αμπάς, θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στη σημερινή πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας καλωσορίζω εγκάρδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εταίρος της Παλαιστίνης στις χρηματοοικονομικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές ε, σχέσεις. Μία ε, Παλαιστίνη που να λειτουργεί σωστά είναι και ηθικό καθήκον για μας. Κύριε Πρόεδρε Αμπάς, αφιερωθήκατε, αφιερώσατε τη ζωή σας στο Παλαιστινιακό στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, στην ελευθερία και χωρίς βία. Ήσασταν από τους αρχιτέκτονες της Ειρηνευτικής Διάσκεψης Μαδρίτης και της Συμφωνίας του Όσλο. Μέχρι σήμερα αποτελείται ορόσημο της συνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Σήμερα η παρουσία σας εδώ, μετά την ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου Ρίβλιν, χτες, είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η βούληση για μια αηφόρο και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης παραμένει ζωντανή. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να εξάρω την ακούραστη εργασία της κυρίας Μογκερίνη, υπάτης εκπροσώπου που παρευρίσκεται σήμερα το πρωί, όπως ήταν παρούσα και χτες το απόγευμα. Καλώς ορίσατε και εσείς κυρία Μογκερίνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο 2015 απεφάθη για ε, μία λύση δύο κρατών βάσει των συνόρων του 1967 με ε, την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών. Σε αυτή τη λύση των δύο κρατών θα πρέπει να υπάρχει ένα Ισραήλ που να ζει με ασφάλεια, το είπα και χτες και το υπογράμμισα, αλλά και μια ανεξάρτητη, δημοκρατική, ε, ε, ζωντανή Παλαιστίνη που να είναι ένα κράτος βιώσιμο με συνοχή και θέλω να το υπογραμμίσω και σήμερα. Και θα πρέπει να ζουν με ασφάλεια χέρι με χέρι, δίπλα-δίπλα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πρώτα να τερματιστεί η βία. Κανένας πολιτικός στόχος δεν δικαιολογεί το τυφλό μίσο την υποδάβλησή του ή το, την τρομοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει και όχι για πρώτη φορά ε, την επέκταση των Ισραηλινών επικισμών καθώς επίσης ε, και την εκτόξευση ρουκετών προς το Ισραήλ από ομάδες ε, μαχητών. Αυτό οδήγησε σε έναν αποκλεισμό της Γάζας που θα πρέπει να λυθεί και το έχουμε ζητήσει και έχουμε ζητήσει και μια συμφιλίωση. Συμφιλίωση μεταξύ των Παλαιστινίων για ε, συγγνώμη, για συνέστηση, ενσυναίσθηση και μεταξύ των Παλαιστινίων αλλά και μεταξύ Πανεστινίων και Ισραηλινών. Αυτό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της συνευτικής διαδικασίας για την οποία εσείς αγωνίζεστε. Σας καλωσορίζω και όλων των συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας δίνω αμέσως με χαρά το λόγο. Παρακαλώ.